Dear colleagues. Συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας. Πριν όμως ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους συναδέλφους να τηρήσουν σιγή για όσα συνέβησαν σήμερα το πρωί στο Ζάβεντον. Thank you very much. Item 9 in our agenda. Το σημείο 9 στην ημερήσια διάταξη ανακοίνωση του Προέδρου για τις συστάσεις των συντονιστών από την 21η Μαρτίου. Οι συστάσεις των συντονιστών έχουν κυκλοφορήσει ηλεκτρονικώς και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα θεωρηθούν εγκεκριμένως. Συνεχίζουμε τώρα με την ψηφοφορία. Πριν ξεκινήσουμε πρέπει να κάνουμε μια επαλήθευση για την έκθεση Νικολάφιτ. Έχουμε έτοιμα για ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία 36, 37 και 38. Και θα πρέπει να βεβαιωθούμε ποιοι είναι υπέρ του αιτήματος αυτού και ποιοι κατά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τα ψήφισαν άπαντες. Όχι. Πέρας της ψηφοφορίας. Το αίτημα απορρίπτεται. Και να ξεκινήσουμε τώρα την ε, ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρα. Εγκρίνεται. Κυρία Ζόμερ, με συγχωρείτε που καθυστέρησα. Δεν έχω την κάρτα μου. θα μπορούσα να ψηφίσω διαγάτας ισχυρός. Άντε εντάξει, αλλά αν μπορεί η βοηθό σας να πάει να φέρει την κάρτα. Ναι, ναι, τρέχει ήδη. Όσο πιο γρήγορα μπορεί παρακαλώ. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. να άπαντες πέρας. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4, συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά αποχές κρίνετε. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία για την 37 υπάρχει προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία του κυρίου Μεκολάσιτς. Αντίρρηση κυρία Ντάλ. Πάνω από τέσσερις. Ψηφίζουμε λοιπόν χωρίς την προφορική τροπολογία σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 40 υπέρ, κατά, αποχές, αγκρίνεται. 41 κατά πίπη, 42 υπέρ, κατά, αποχές, Αγκρίνεται Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61, συμβατή, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 62, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 74 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 79 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική και η συνάδελφος Σόμαρα έχει πλέον την κάρτα της. Εψήφισαν άπαντες πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ψηφοφορία για το ψήφισμα για την υποχρεωτική ένδειξη γεωγραφικής προέλευσης και ορισμένων τροφίμων, τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρα τη ψηφοφορία ψήφισαν άπαντες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, ε, τροπολογία 39 σε δύο τμήματα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 38 σε δύο τμήματα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει επειδή το πρώτο τμήμα απορρίφθηκε. Τροπολογία 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη. 41, ε, 42 και 43 πανομοιότυπες ε, σε μπλοκ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 45 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Πέρας με μία ψήφο διαφορά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 47 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49. Μαζί με την 50 πανομοιότυπες υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 52. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. κατά έλεγχος. Εψήφισαν άπαντες πέρας. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει 54 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίβεται, 57 υπέρ κατά αποχές έλεγχος Πέρας. Εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 65 σε δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68. Απορχές απορρίπτεται. 79. 69, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έλεγχος. Avete votato tutti? Εψήφισαν άπαντες, πέρας εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 72 κατά, αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 74 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υπέρ. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα 75, 76 και 77 που είναι πανομοιότυπες από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σε δύο τμήματα τα 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα Με συγχωρείτε, η τροπολογία 78 κατέπεσε, διότι εγκρίναμε την 81. Οπότε καταπίπτει και δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε την 78, ούτε την 79. Πρέπει να ψηφίσουμε την 80, επί της οποίας υπάρχει προφορική τροπολογία του κυρίου Φιέλνερ. Έχετε κάποια αντίρρηση για την προφορική τροπολογία. Εάν όχι, να ψηφίσουμε την 80 όπως τροποποιήθηκε με την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. 83 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Avete votato tutti? Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Εγκρίνεται. πέντε. υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Σε δύο τμήματα. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει. 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 89 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 94 απορρίπτεται. 91 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το 92 δεν θα ψηφιστεί. Τροπολογία 97. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 103 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 114 Γκαρντίνη Τσίριο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 111. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Εκατόν δεκαοκτώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. Έλεγχος. 118. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 115. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 120. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 113. Υπέρ. Κατά αποχές, έλεγχος. Πολύ λίγοι σηκώνουν τα χέρια τους. Εψήφισαν άπαντες πέρας. Πέρας, εγκρίνατε. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 119. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 106. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Αγκρίνεται. Εκατόν επτά. Επειδή 116 καταπίπτει. 107. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 117 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 108 υπέρ, κατά, να συγχωρείτε. 108 καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε η 74. Τροπολογία 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 112. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. Πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται με μια ψήφο διαφορά. Δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί είστε διχασμένοι στις πολιτικές ομάδες, οπότε γι' αυτό χρειάζεται παλήθευση. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Εψήφισαν άπαντες πέρας. Απορρίπτεται. Μπορούν οι σοσιαλιστές να σηκώνουν τα χέρια τους. Ψηφίζουμε την ε, τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18. καταπίπτει. 17. Υπέρ της 17. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά έλεγχος. Εψήφισαν άπαντες πέρας. Εγκρίνεται. Δεκαεννέα. υπέρ, κατά, έλεγχος. Τα πάντε πέρας εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εψήφισαν άπαντες. Απορρίπτεται. 24 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα το σχέδιο ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία προφανώς. Υπέρ. Άρχια τη ψηφοφορία. Εψήψαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τις ψηφοφορίες μας. Παρόλο που ε, έλαβε χώρα και άλλη τρομοκρατική μάλλον επίθεση στο μετρό. Περνάμε στην ψηφοφορία για την επιδημία του ιού του Ζίκα. Ξεκινάμε με την τροπολογία 17. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Avete votato tutti, Il voto è chiuso. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Συμβατή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 της Επιτροπής ΔΕΒΕ. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 25. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 της Επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 της ΔΕΒΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 31 καταπίπτει, τροπολογία 32 τώρα, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 34 τροπολογία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 της Επιτροπής ΔΕΒΕ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 για την παραγράφο 18α9 της Επιτροπής των Γυναικών. Α, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 38. Avete votato tutti, il voto è chiuso, approvato. Emendamento 39. Chi è a favore? Τροπολογία 39. Ποιος είναι υπέρ? Με 38 εγκρίθηκε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 40. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 δεύτερο τμήμα που είναι συμβατό. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 της ΔΕΒΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 4 και τροπολογία 47 πανομοιότυπες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 53 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 48 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στι ιδεολογικέ σκέψη τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε την τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1 της Επιτροπής Γυναικών. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δύο της Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 9. Τα υπόλοιπα κατέπεσαν υπέρ, παρακαλώ. Του δεύτερου τμήματος 9 κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας παρακαλώ. Εγκρίνεται. The next vote will be on η επόμενη ψηφοφορία αφορά τη διαδικασία αντίρρησης. Α, συγγνώμη, κυρία Ντελαέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για την επόμενη ψηφοφορία θα ήθελα να πω ότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε τις αντιρρήσεις. Ε, δεν αρκεί να είναι κανείς υπέρ ή κατά όπως ε, μας ζητά σήμερα να ψηφίσουμε η αντίρρηση. ζητα ουσιαστικά ζητά η αντίρρηση από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ανανεώσει την άδεια και να υποβάλει νέα πρόταση. Θα πρέπει να έχουμε μια μέσο και μακροπρόθεσμη προοπτική, κυρίω για του καταναλωτέ που θέλουν υγιεινά τρόφιμα, αλλά και για του γεωργού, που είναι οι χρήστε κυρίω αυτή τη ουσία και βιώνουν μια σοβαρή κρίση. Ελπίζω μέχρι την Ολομέλη να συνεργαστούμε με του συναδέλφου και να διατυπώσουμε τροπολογίε με επικοδομητικά και χειρά μηνύματα προ τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι αρμόδια για το θέμα αυτό. Σα ευχαριστώ. Μάλιστα. Πρώτα θα ψηφίσουμε το, το σχέδιο ψηφίσματος το κοινό πολλών ομάδων ηλεκτρονικά. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτει το εναλλακτικό σχέδιο ψηφίσματος της ΕΝΕΦ, της Ομάδας των Εθνών και των Ελευθεριών. Και ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες μας. Παρακαλώ, αν κάποιος θέλει να βγει από την αίθουσα, αθόρυβα παρακαλώ και γρήγορα. Σε ένα λεπτό περνάμε στην επόμενη, στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Eh, oppure faccio uscire qualcosa a per Αγαπητοί συνάδελφοι, συνάδελφοι, νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση είναι να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Και μετά θα σας πρότεινα να περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημέρας της διάταξης, Επιστολή Ένβη στο Μοντρεάλ. Στον Νικάο, ΚΑΙΠ 10. Σε αυτό λοιπόν το σημείο θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της ε, αντιπροσωπείας, η κυρία Γκέρλινγκ, για να μας παρουσιάσει την, ε, τι έγινε και μετά θα το συζητήσουμε. Κύριε Γκέρλιν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δυστυχώ δεν έχω μαζί τι σημειώσει μου και πολύ σα ζητώ συγγνώμη. Λυπάμαι, αλλά σήμερα το πρωί ήρθα κατευθείαν εδώ και προσπαθεί να τη φέρει τώρα ο, η βοηθός μου. Θα σας τα πω όπως το θυμάμαι. Όλοι λάβατε την γραπτή έκθεση. σε ό,τι αφορά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας. Όπως ξέρετε ήταν μια αποστολή η οποία διοργανώθηκε υπό δύσκολου όρους και αυτό γιατί το Κοινοβούλιο δεν έλαβε την έγκριση να μεταδεί στην συνάντηση ΚΑΚ. Και έτσι έχουμε την αίσθηση, είχαμε την αίσθηση ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα, αλλά είναι σαφές ότι πρόκειται για μια πολύ τεχνική συνάντηση και ως εκ τούτου το γεγονός ότι δεν συμμετείχαμε στις ε, ολομέλειες τελικά και χάρη στην εξαιρετική εργασία της γραμματείας μας και της ε, αντιπροσωπείας της Κομισιόν θεωρώ ότι καταφέραμε στο Μοντρεάλ να σημειώσουμε τελικά σημαντική πρόοδο τις ημέρες αυτές που είχαμε εκεί. Τι κάναμε λοιπόν, διοργανώσαμε μία σειρά διμερών συναντήσεων εκτός ε, της, των επίσημων συναντήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι προφανώς συμμετείχαν πολύ σημαντικά άτομα εκεί, τα άτομα με τα οποία ουσιαστικά θα έπρεπε να συνομιλήσουμε, με τα οποία θα έπρεπε να συνομιλήσουμε για τους μηχανισμούς της αγοράς. Ως εκ τούτου, αρχικά διοργανώθηκαν κάποιες συναντήσεις με τις ΜΚΟ, πολύ χρήσιμες και ωφέλιμες εν γέννη. Έγιναν συναντήσεις με διάφορες άλλες οργανώσεις και τις ε, ομάδες και ενώσεις ε, αρχών ε, του αεροδρομίου, τις αεροπορικές γραμμές στα πλαίσια της ΙΑΤ και με διάφορες επίσης χώρες διμερείς συναντήσεις διοργανώθηκαν. Έλειψαν κάποιες σημαντικές χώρες. Η πιο σημαντική χώρα με την οποία δεν καταφέραμε να συνδεθούμε ήταν η Κίνα. Νομίζω εν μέρει επειδή ήταν και το... οι εορτασμοί του νέου έτους ε, για τους Κινέζους. Και αυτό είναι... ήταν κρίμα γιατί προφανώς και οι Κινέζοι παίζουν μεγάλο ρόλο και δεν καταφέραμε να συναντηθούμε μαζί τους. Καταφέραμε να συναντηθούμε και με άλλους ε, εταίρους ε, και η πιο βασική ήταν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αυτούς συναντηθήκαμε και ξεχωριστά και όλοι μαζί. Ήταν σημαντικό αυτό, γιατί προφανώς θα συνεργαστούμε μαζί στις επόμενες συναντήσεις και στη συνέλευση. Επίσης, ε, χρήσιμες συναντήσεις και με την χώρα υποδοχής των Καναδά, γιατί προφανώς και έχουν ε, πολλά και βάσιμα στοιχεία για να μας δώσουν και κυρίως για τις ΗΠΑ. Άρα, δεν ξεκίνησε καλά η συνάντηση και υπήρχε γενικά ένα νέφος, μια ομίχλη. Αλλά γενικά νομίζω ότι κατέληξαν πιο θετικά, πιο αισιόδοξα οι συναντήσεις. Ήταν σαφές το μήνυμά μας, αλλά παράλληλα δεν έπρεπε να το θέσουμε το μήνυμα με τέτοιο τρόπο. ώστε να θεωρηθεί όπως πολλοί μας είπαν ως ε, κάτι, ως μία έκκληση να σταματήσουμε το χρόνο και να επανέλθουμε σε αυτά που ίσχυαν στα τέλη του προηγούμενου έτους. Ήταν σαφές λοιπόν ότι δεν ε, απειλούσαμε τους υπόλοιπους και δεν τους λέγαμε ουσιαστικά, δεν τους υπαγορεύαμε ότι ο ευρωπαϊκός τρόπος ήταν ο μοναδικός τρόπος που θα έπρεπε να ακολουθήσουν. Ήμασταν αρκετά διπλωματικοί. Ήταν αρκετά περίεργη η θέση μας. Καταφέραμε να συναντηθούμε με τον πρόεδρο της ΕΚΑΟ και εγώ προσωπικά είχα την αίσθηση ότι ήταν πραγματικά πολύ διαφωτιστική αυτή η συνάντηση. Ο πρόεδρος του ΙΚΑΟ μας έθεσε τους προσωπικούς στόχους του για την ε, ολοκλήρωση ενός μηχανισμού μέχρι το Σεπτέμβριο σε ό,τι αφορά τους στόχους για τον άνθρακα, τους οποίους εμείς ενδεχομένως ε, θεωρούσαμε ότι ήταν πιο χαμηλοί σε σχέση με αυτά που είχαν υποσχεθεί, αλλά ήταν σημαντικό το ότι είχαν καταφέρει να συμφωνήσουν από αυτόν. Ήμασταν λοιπόν και τα ικανοποιημένοι εν τέλει, τον συγχαρήκαμε και τονίσαμε ότι θα θέλαμε να συμμετέχουμε στην επόμενη συνάντηση τον Μάιο δεσμεύτηκε επί της αρχής ε, ο πρόεδρος ότι δεν θα είχε αντίρρηση να, συμμετέχει για την προσωπία του Κοινοβουλίου στην βασική συνάντηση το Μάιο. Αυτά λοιπόν ως προς τα επιτέγματα των δύο ημερών. Ελπίζω. Και πολύ σας ζητώ συγγνώμη, δεν έχω τις ε, σημειώσεις μου μαζί, όπως σας είπα και στην αρχή. Αν έχετε ωστόσο ερωτήσεις, θα χαρώ να τις απαντήσω. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Γκέρλινγκ για την προσπάθειά σας να τα θυμηθείτε όλα αυτά. Δεν ξέρω αν έχουμε μαζί μας συναδέλφους που συμμετείχαν. Ο κύριος Μπελέτ, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω αυτά που εξαιρετικά μας παρουσίασε η κυρία Γκέρλινγκ στην ενημέρωσή της να τη συγχαρώ για την ε, εξαιρετική της προέδρια της αντιπροσωπείας αυτής και την γραμματεία να συγχαρώ. Δεν ήταν καθόλου εύκολη η εργασία τους. Το αντιλαμβανόμαστε. Σας ευχαριστούμε. Και να συγχαρούμε και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξαιρετική συνεργασία και μαζί τους στον Καναδά. Ήδη η κυρία Ντέρλινγκ μας μίλησε για το πρότυπο για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό αποτέλεσε ασφαλώς μια πρόοδος, αλλά εκ παραλλήλου ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν ήταν και φιλόδοξη τελικά η απόφαση σε σχέση με τον στόχο που ετέθησε. Ελπίζω μεσοπρόθεσμα να περάσει από αναθεώρηση. Και το δεύτερο θέμα το οποίο επίσης αναφέρε η κυρία Γκέρλινγκ, αυτός ο μηχανισμός για την παγκόσμια αγορά, ο οποίος βρίσκεται υπό κατασκευή. Ελπίζουμε να εγκριθεί το Μάιο, να εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ξέρουμε ότι όλοι έχουμε ανάμεκτα συναισθήματα σε σχέση με αυτά που πλέον έχουμε μπροστά μας στο τραπέζι διαπραγματεύσεων στον ΙΚΑΟ γιατί δεν μιλάμε για ένα ETS, ένα μηχανισμό εκπομπή εμπορία ε, ρήπων ή ε, έστω με μια εναλλακτική αυτού αλλά ένα μηχανισμό αντιστάθμισης, ε, offset, που περιλαμβάνει πολλές εξαιρέσεις και απαλλαγές για πολλά κράτη, για πολλές χώρες. Ούτε αυτό μας ικανοποιεί και ο διάολος από ό,τι ξέρετε κρύβεται στις λεπτομέρειες. Αυτό που έχουμε λοιπόν μπροστά μας μας προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα. Η Julie Γκέρλινγκ αναφέρθηκε στο μηχανισμό ε, Stop the Clock για να ε, γυρίσουμε πίσω το χρόνο, για να σταματήσουμε το χρόνο μάλλον για τα όσα θα ισχύουν μέχρι τα τέλη του έτους. Και πρόσφατα παρατηρήσαμε ότι η διεθνής ε, αεροπορία σύμφωνα με τις πρόσφατες ερευνές, ε, ε, μέχρι το 2050 θα έχει καταστεί βασικός, ε, βασική πηγή εκπομπής τέτοιων αερίων. 20 30% μέχρι το 2050. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ευθύνη που βαρύνει τη διεθνή αεροπορία τα επόμενα χρόνια είναι μεγάλη και θα πρέπει το έργο τη και τα καθήκοντά τη να εκπληρωθούν με πιο σοβαρό τρόπο. Ελπίζω λοιπόν τουλάχιστον να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε για ένα μηχανισμό αντιστάθμιση, αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό να είναι και το τελικό καταληκτικό σύστημα, ο τελικό μα και απότερος στόχος. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν μια μεγάλη πρόκληση σε ό,τι αφορά το μηχανισμό αυτό στο the clock ε, θα εγκριθεί αυτός ο μηχανισμός. Δεν είναι ιδανικό σε καμία περίπτωση, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα. Αν εγκριθεί, θα θέλαμε να εγκριθεί και στο Κοινοβούλιο, αλλά αυτό είναι μια προκαταρτική σκέψη και φυσικά όλα θα εξαρτηθούν και θα πρέπει να υπάρξει και ένας ταχύτατος μηχανισμός αναθεώρησης. Μόνο έτσι νομίζω ότι θα καταφέρουμε να εγκρίνουμε και να συμφωνήσουμε στο μηχανισμό αυτό, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση οπωσδήποτε στο Κοινοβούλιο και θα δούμε και πώς θα δημορφωθεί η κατάσταση μέχρι το τέλη του έτους. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ. Κανείς άλλος Ο κύριος Λίζα και ο κύριος Γκρότα. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και τον συναδέλφου που περάσαν όλο αυτό το τραπατσάρισμα γιατί ήταν δύσκολη αυτή η αντιπροσωπεία. Δεν ήταν και σαφές κατά πόσον θα γινόντουσαν και σωστές συζητήσεις ε εξ αρχής, γιατί στην αρχή οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιοι του ΙΚΑΟ δεν θέλαν καν να δεχτούν την αντιπροσωπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε όμως τους συναδέλφους που παρόλα αυτά πήγαν, μετέβησαν στο Μοντρεάλ και τελικά κατάφεραν να κάνουν και ωφέλιμες και χρήσιμες συναντήσεις. Ο σκοπός που έχουμε όλοι μας είναι να βρούμε μία παγκόσμια λύση για τις εκπομπές από την αεροπορία. Και δυστυχώς ε, διαπιστώνουμε ότι στις διεθνείς διαπραγματεύσεις τα πράγματα πηγαίνουν ε, πάντα αργά. Και ούτε και το Παρίσι πρέπει να παραδεχτούμε ήταν τόσο ε, σημαντικό επίτευγμα για να θεωρήσουμε τα έχουν τα προβλήματα. Αλλά δυστυχώς και στον ΙΚΑ τα πράγματα πηγαίνουν ακόμα πιο αργά και αδύναμα από τη σε σχέση με τις διεθνείς συναντήσεις. Από το 2020 και μετά το σκοπός είναι να υπάρχει μια ουδέτερη ανάπτυξη σε ό,τι αφορά τις εκπομπές, άρα δεν μιλάμε καθόλου για μείωση των εκπομπών. Δεν τίθεται καν τέτοιο θέμα. Πρώτο πρόβλημα θεωρώ είναι αυτό. Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό γιατί και η ίδια, ο ίδιος ο οικονομικός ε, κλάδος, η ΙΑΤΑ, έχει ήδη θέσει από μόνο του το στόχο της μείωση κατά 50% μέχρι το 2050 των εκπομπών. Είναι θέμα που πρέπει να το δείξουμε αυτό. Στου υπεύθυνου του ΙΚΑΟ, του ουσιαστικά δηλαδή ο ίδιο οικονομικό κλάδο οι επιχειρήσεις είναι πιο φιλόδοξες από ότι οι ενώσει και οργανώσεις. Carbon Neutral Growth, ε, ανάπτυξη με ουδέτερη, με ουδέτερες εκπομπές άνθρακα. Μιλάμε για αντισταθμίσεις των αεροπορικών εταιριών προς τις άλλες οικονομικούς φορείς οι οποίοι κάνουν προσπάθειες και καταβάλουν προσπάθειες. Οι υπεύθυνοι του ΙΚΑΟ θεωρούν ότι μπορεί να πετύχουμε συμφωνία μόνο αν ε, αποδυναμωθεί εκ νέου αυτός ο στόχος για την ε, ανάπτυξη με ουδέτερε εκπομπέ ανθρακά, με με μηδενικές, ε, με μηδενική αύξηση του άνθρακα, των εκπομπών του άνθρακα. Άλλες χώρες τώρα, όπως η Κίνα, θα ενταχθούν στις όλες τις συμφωνίες από το 2024 και μετά. Αυτό αποτελεί ένα επιπλέον πρόβλημα. Στο Παρίσι ε, συμφωνήσαμε ότι το τριπλό σίτι σημαίνει ότι όταν ε, χώρες όπως η Κίνα και οι χώρες του τυπικού του υποανάπτυξη ε, έχουν περιθώριο να μην έχουν τέτοιους στόχους και προσωπικά να μπορούν να αυξήσουν τις εκπομπές τους, αυτό θα πρέπει να αντισταθμίζεται από περαιτέρω μείωση των εκπομπών από τις εκβιομηχανισμένες ε, αναπτυγμένες χώρες. Ε, αυτό δεν ε, διευκρινίζεται όμως στον ΙΚΑΟ Και γι' αυτό πιστεύω λοιπόν ότι τους επόμενους μήνες θα πρέπει να καταβάλουμε επιπλέον προσπάθειες και θα το απέφτεινα αυτό ως έκκληση και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, αν είναι παρούσα και προς τα κράτη-μέλη που κάνουν διαπραγμάτευση άμεσα στον ΙΚΑΟ. Να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε πιο φιλοδόξους τους στόχους μας. Ε, φέτος δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία η οποία να είναι και έτοιμη προ επικύρωση μέσα στο έτος. Θα υπάρξει μόνο μια πολιτική δέσμευση επί τη οποία θα συνεχίσουν οι εργασίες. Θα πρέπει να υπάρχει και μια ρήτρα αναθεώρηση τουλάχιστον για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το στόχο που έχει θέσει ο ίδιο ο κλάδο, το μείον 50% μέχρι το 2050. Αυτό που θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε εμεί σε πιο βραχυπρόθεσμο επίπεδο είναι το τι θα κάνουμε με την αεροπορία και τι αεροπορικέ μεταφορέ στην Ένωση ε, άμεσα θέλαμε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να συμπεριληφθούν στο ETS όλες οι πτήσεις που προσγειώνονται στην Ευρώπη και προκειμένου μια πτήση από την Αθήνα στο Λονδίνο, από τη Φραγκφούρτη στη Ρώμη, να καλύπτονται, αλλά όχι οι διπηρετικές ε, Ε. Αλλά ο στόχο είναι και αυτός ο δυνάμος. Ο 10% στη Χαλιβουργία, για παράδειγμα, είναι πολύ πιο υψηλή, στόχη. Δεν θέλω να πω ότι δεν έχει προβλήματα και ο αεροπορικός κλάδος, αλλά σε σύγκριση με τη Χαλιβουργία, ας πούμε, είναι πιο ε, λίγα τα προβλήματα. Η Χαλιβουργία αγωνίζεται να επιβιώσει. Στο ETS ε για τους ε, τομείς ε, που δεν ε, εμπλέκεται η διαρροή άνθρακα έχουμε 100% προσαρμογή, μόνο 15% όμως για τις πτήσεις. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Μέσω μέχρι τον Σεπτέμβριο, γιατί στην συζήτηση για την αεροπορία, γίνεται μια συζήτηση για την διαρροή άνθρακα, γίνεται και μια συζήτηση σε ό,τι αφορά α, ε, τις πτήσεις α, ε, μέσω Μεσανατολής, υπάρχει και το θέμα της διαρροής άνθρακας ε, στην Χαλιβουργία και σε άλλες υψηλής έντασης βιομηχανίες. Το θέμα φυσικά είναι ότι υπάρχει και το θέμα ε, της ε, αντικατάστασης φυσικά της παραγωγής της χαλιβουργίας με εισαγωγές. Αλλά δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε μία πτήση από την Αθήνα στο Λονδίνο, από την Φραγκφούρτη στο, στη Ρώμη. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε σε ό,τι αφορά και τις διπυρωτικές ε, πτήσεις. Να μην δημιουργήσουμε την εντύπωση ότι εντάξει, μας κάνουν μας κάνει οποιαδήποτε λύση, ακόμα και αν δεν έχει ουσιαστική βελτίωση και επίπτωση στο Κοινοβούλιο. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα κοιτάξουμε στις διαπραγματεύσεις μας στα πλαίσια του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τον κύριο, και λέει και ο κύριος Δεκρότα, για να ευχαριστήσω την προσωπία που μου ε, πήγε στον ΙΚΑΟ. Ήταν πραγματικά ε, επικίνδυνη αποστολή, Mission Impossible, αυτή που έλαβε χώρα εκεί, αλλά πραγματικά έκανε πολύ καλά συνομιλίες, πέτυχε πολύ καλά αποτελέσματα και έθεσε το μήνυμα και το σήμα ότι είμαστε και παρακολουθούμε την κατάσταση και ότι είναι δικό μας καθήκον να παρακολουθούμε την κατάσταση και να μην αρκούμαστε ε, σε αυτά που συζητιούνται. Γιατί εμείς είμαστε ο νομοθέτης, εμείς πρέπει να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και εμείς ε, θα πρέπει να τα παρουσιάσουμε αυτά και στους πολίτες. Δεν εξαρτάται αυτό από ε, κάθε υπάλληλο στην Κομισιόν για την διαρροή άνθρακα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα, το είπε και ο κύριος Λίζε, σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του ETS, να υπάρχει μια στρατηγική γιατί υπάρχουν ε, τομείς που έχουν ειδικό ρόλο, αλλά όλοι οι οικονομικοί κλάδοι είναι μέσα στη διεθνή ανταγωνισμό. Και γι' αυτό λοιπόν ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να πετύχουμε ένα σωστό συμβιβασμό στην τελική ανάλυση, τον οποίο να υποστηρίξει και μια μεγάλη πλειοψηφία Γιατί μόνο έτσι θα πετύχουμε αποτελέσματα, όχι με μια πλειοψηφία οριακή εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντο, για να δείξουμε ότι είμαστε σοβαροί σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντο και ότι κάθε τομέα θα πρέπει να συμμετέχει και να κάνει τι αντίστοιχε προσπάθειε. Ξέρω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα σε διεθνέ επίπεδο, αλλά. Πώς να εξηγήσω τα πράγματα αυτά ε, σε οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε εκπροσώπους της Χαλιβουργίας για παράδειγμα ότι κοιτάξτε σε εσά ε, είμαστε αυστηροί και σε εσά και στην ε, παραγωγή τσιμέντου αλλά ξέρετε στην αεροπορία είμαστε λίγο πιο ελαστικοί. Δεν γίνεται. Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες και αποφασίσαμε λοιπόν να συνεχίσουμε τη συμμετοχή μας στις περιπτώσεις συναντήσεις και συνεδρίες του ΙΚΑΟ ως Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε συνάδελφοι και θα πρέπει να καταφέρουμε να σχηματίσουμε ένα συμβιβασμό, μια γραμμή συμβιβασμού, την οποία να υποστηρίξουν όσο πιο πολλοί συνάδελφοι γίνεται. Thank you very much. I don't know if... Ευχαριστώ. Δεν ξέρω κάποιος άλλος συνάδελφος ενδιαφέρεται να μιλήσει. Όχι. Οπότε μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό της ημίρησης διάταξης και να περάσουμε στο επόμενο, το τελευταίο για σήμερα. Ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υγειονομική περιθέψη των προσφύγων. Θα θυμάστε ότι μια πολιτική ομάδα κατέθεσε σχετικό αίτημα και θα δώσω το λόγο πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστώντας την που ε, δίνει το παρόν ακόμη και σήμερα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον εκπρόσωπό της για μια εισαγωγή και θα ακολουθεί η συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής. Η κυρία Ιζαμπέλ Ντελαμάτα Μπαράνκο. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Από την αρχή αυτής της έκτακτης κατάστασης με τις μαζικές εισορές προσφύγων και μεταναστών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δραστηριοποιήθηκε σε όλα τα μέτωπα, ακόμη και στην υγεία. Και μάλιστα έχουμε ε, μια ένα συντονισμό των δραστηριοτήτων στην Επιτροπή Υγείας ε, προκειμένου να χορηγούμε εμβόλια, να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν για διαγωνισμούς και προμήθειες ε, και να έχουμε το σύστημα έγκαιρης ε, προειδοποίησης και επαγρύπνησης για τις λοιμώδεις νόσους σε συντονισμό με τα εθνικά σημεία επαφής και τις αρχές για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες και επίσης ε, να λαμβάνουμε υπόψη την υγειονομική κατάσταση των προσφύγων. Συμβάλλουμε στην καλύτερη τύλιψη του γεγονότο ότι οι μαζικέ ροές προσφύγων και μεταναστών δεν αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία, ούτε για του αφιχθέντε, ούτε για τον πληθυσμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η παρακολούθηση πιθανών απειλών γίνεται με βάση το σύστημα επαγρύπνηση και είμαστε έτοιμοι να λάβουμε και κατεπήγοντα μέτρα αν εντοπιστούν ιδιαίτερε ανάγκε. Από κοινού με την Διεθνή Οργανισμό για την Μετανάστευση και με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη των Νόσων ετοιμάζουμε ένα νέο ε, εργαλείο για την αποτίμηση της υγειονομικής κατάστασης των προσφύγων. Μάλιστα έχουμε ένα εγχειρίδιο που ε, υπάρχει και στα αραβικά και σε πολλές γλώσσες το σχετικό εγχειρίδιο για το νοσηλευτικό προσωπικό. Μάλιστα έχουμε και ένα περιοδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα και θα το επεκτείνουμε στην Ιταλία, Σλοβενία και Κροατία. Θα υπάρχει και ηλεκτρονικά και γράφος για να εξασφαλίσουμε ανταλλαγή πληροφοριών με τις χώρες προορισμού. Επίσης ε, έχουμε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα HELP για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να αντέξουν τις ε, μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές και τις υγειονομικές επιλές. Επίσης έχουμε τέσσερα πλέον προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν για ένα χρόνο, ξεκινώντας από τις 3 Ιανουαρίου του 2016. Είναι συμπληρωματικά αυτά τα σχέδια και ε, προβλέπουν πρωτόκολλα, κατευθυντήριες γραμμές ε, και μέσα συντονισμού. Επίσης ε, συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Ιατρικό Σώμα για την υγειονομική περίθαλψη. Ε, βέβαια, μας ενδιαφέρει ολοκληρωμένη προσέγγιση και το σχέδιο εργασίας του 2016 ε, θα αφιερώσει 7,5 εκατομμύρια ευρώ σε δραστηριότητες και βέλτιστες πρακτικές για μοντέλα υγείας ε, για και την ένταξη των προσφύγων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχική υγεία. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 4 Μαρτίου και πριν το καλοκαίρι θα έχουμε δύο διαγωνισμούς και για την κατάρτιση από κοινού με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας θα συμπληρώσουμε αυτά τα μοντέλα με το μοντέλο για τις λοιμώδεις νόσους και την ψυχική υγεία. Και κυρίως ε, πρόκειται για προγράμματα για τους ε, μεθοριοφύλακες ε, και το νοσηλευτικό προσεκτικό. Και κυρίως στις χώρες της, νότια, της Νότιας Ευρώπης. Να, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ειδικέ ανάγκες των προσφύγων. Έχουμε και την ομάδα εργασίας ε, για το νοσηλευτικό προσωπικό που θα ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Υγειονομικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι μια περίληψη των δραστηριοτήτων που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν έχουμε ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Κυρία... Κυρία Μπέρντερ. Ναι, ίσως δεν άκουσα, αλλά είπατε πώς ε, μπορούν οι οικογένειες να παραμένουν ενωμένε, διότι αν κάποιος στάσει και χρειάζεται περίφαλψη, εισαγωγή σε νοσοκομείο, δεν χωρίζονται οι οικογένειες έτσι. Πώς φροντίζετε να διατηρήσουν την επαφή μεταξύ τους οι οικογένειες εάν χρειάζονται ιατρική φροντίδα και τα άλλα μέλη της οικογένειας βρίσκονται αλλού. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αρμόδια για, αυτήν την, ε, για αυτόν τον τομέα. Ο οργανισμός η υγειονομικής περίθαλψη και η διοργάνωση των θεμάτων αυτών είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εδώ όμω δεν μιλάμε για υγειονομική περίθαλψη, μιλάμε για κοινωνική πρόνοια και την βοήθεια προς τις οικογένειες. Αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συγχωρείτε πολύ, αλλά δεν έχω αρμοδιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ήταν το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Η επόμενη συνεδρίασή μας είναι στις 18-19 Απριλίου και μπορούμε να κηρύξουμε εδώ τη λήξη της σημερινή μας περίεργης συνεδρίασης λόγω των δυσκολιών έξω. Ευχαριστούμε πολύ και θα σας δώσω την επόμενη συνεδρίαση.